Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Σε συμφωνία με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, και επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων που περιμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, θα σας δώσω τα αποτελέσματα αυτά. Μετά, μόνο μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει γίνει η πλήρη συγκρότηση σε σώμα του Κοινοβουλίου. Κάνω λοιπόν αυτή την ανακοίνωση. Και οι 14 έχουν εκλεγεί. Η σειρά είναι, είναι η σειρά που, προβαδίσματος που ακολουθείται μετά την ε, εκλογή τους. Σας λέω λοιπόν τα αποτελέσματα με τη σειρά των ψήφων. 672 ψήφοι. 17 άκυρες ψήφοι. Έγκυρα ψηφοδέλτια 655. Έλαβον Γιάννη Πιτέλα 319 ψήφους. Μικέλ Άγχελ Μαρτίνες 295 Άννη Ποδηματά 281 281 ψήφους Αλέχο Βίδαλ Κουάδρας 269 Γεώργιος Παπαστάμκος 248. Ρομπέρτα Αντζελίλη. 246. Ότμαρ Κάρας. 244. Έντουαρτ Μακμίλαν Σκότ. 239. Ιζαμπέλ Ντυρό, 238. Αλεξάνδρ Άλβαρο. 235. Ράινερ Βίλαντ 230 Όλτριχ Φλάσακ 223 Γιάσεκ Ποσαζιέβιτς 206 και Λάσλο Σουριάν 188 Όλοι οι υποψήφοι λοιπόν έχουν εκλεγεί και μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν ως εκλεγμένοι αντιπρόεδροι. Θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος δεν δέχεται την εκλογή του στο αξίωμα του Αντιπροέδρου μεταξύ των υποψηφίων, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορώ λοιπόν να συγχαρώ όλους τους εκλεγμένους Αντιπροέδρους. Κυρίες και κύριοι, η σύσταση του Προεδρείου είναι δεδομένη λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει στη συνέχεια η σειρά των συγχαρητήριων και τώρα θέλω να δώσω το λόγο αμέσως στον πρόεδρο Μπαρόζο.